θα ήθελα να αρχίσουμε, σας παρακαλώ. Ε, θα περάσουμε στο σημείο 2, ε, έγκριση της μέσης διάταξης. Το σχέδιο το πήρατε στις 24 Μαΐου. I would like to Sorry. Application of Rule 100, sir. No, but I will just, I, I will inform them. Yeah, yeah, but, but we will be. I would like to propose that. Θα ήθελα να προτείνω και υπό το φως που έγινε στη σύσκεψη των συντονιστών, θα σε ενημερώσω βέβαια γι' αυτό, σε λίγο. Θα πρότεινα λοιπόν να μην κάνουμε τη συζήτηση που στο σημείο 6 για την εφαρμογή του άρθρου 130 του κανονισμού. Σχετίζεται με την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης του κυρίου Σαμπον Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια για ποιο λόγο το προτείνω θα σας παρουσιάσω συνολικά τι προτάσει των συντονιστών και τότε θα σα εξηγήσω. Αν δεν έχετε ένσταση και αν δεν ζητάτε κάποια τροποποίηση, θεωρείται εγκεκριμένη μερίσια διάταξη χωρί το σημείο 6, όπως σα πρότεινα μόλι τώρα. Σημείο 3, ανακοινώσει τη Προέδρου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ενημερώσω πώς ε, αποφάσισε το ΕΛΚ, πώς ε, για την ε, γνωμοδότηση από την ΑΦΚΟ προ την ΑΦΕΤ ε, για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνα. Είναι η ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλία θα ανατεθεί ο ρόλο. του εισηγητή στον David Μακάλιστερ από το ΕΛΚ επίση. Στο μεταξύ έχουμε λάβει δύο προτάσεις ψηφίσματος και συμφωνήσαμε ότι θα ακολουθηθεί η γραπτή διαδικασία και για τις δύο προτάσεις εκτός και αν ζητηθεί συζήτηση δεν έγινε κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα δοθεί συνέχεια. Σοφή Μοντέλ για τη διαφάνεια, για, τη, για το λόμπινγκ από πολυεθνικές και δεύτερον άρθρο 150 της ε, Συνθήκης για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δοθεί συνέχεια λοιπόν στις δύο αυτές προτάσεις. Σημείο 4. Νόσεις για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Ε, ε δεν δώσαν για, τις, για εκθέσεις, ούτε και διορίστηκαν οι συγητές μιλήσαμε για τη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση Σέμφλιν για τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών και από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη συζήτηση που έγινε ε, εκτεταμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μη κυβερνητικέ οργανώσει, επίση όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποφασίστηκε λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην δοθεί συνέχεια και ο Φραν Τίμερμαν, ο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, θα έρθει πριν ε, τι καλοκαιρινέ διακοπέ για να μιλήσουμε μόνο, όχι μόνο για τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Θα φτιάξουμε ένα κατάλογο με διάφορα ζητήματα και θα ήθελα να συμβάλλετε κι εσείς και θα ε, οργανώσουμε μια συζήτηση μαζί του. Για τις αποστολές, η διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε την πρόταση της ΑΦΚΟ για τον Καναδά το, για το Σεπτέμβρη ήταν αυτή η αποστολή. Ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο Σούλτς, προσπάθησα να το εξηγήσω και να αιτιολογήσω διότι ε, αυτή η απόρρευση της διάσκεψης των Πρόεδρων ε, δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς στην ε, ΑΦΚΟ. Και εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα αναθεωρηθεί η απόφαση. Προσπαθήσαμε και θα ξαναπροσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων επίσης. Συζητήσαμε για το χρονοδιάγραμμα για την επίσκεψη στην Πολωνία είχαμε προβλήματα να προσδιορίσουμε μία ημερομηνία στα πλαίσια αυτών που προβλέπει το Κοινοβούλιο γιατί πρέπει και οι επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου στην Πολωνία να είναι διαθέσιμες ε, όταν θα μεταβούμε στη χώρα και θα πρέπει να βρούμε εκτός ε, φυσιολογικών σλότ, εκτός χρονοδιάγραμματος του Κοινοβουλίου, να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε με μία γλώσσα μόνο, να μην έχουμε μετάφραση. Το σημαντικό είναι ε, να βρούμε μία ημερομηνία όπου θα ε, συζητήσουμε με εκπροσώπους και των δύο επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου και των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου. Για το σημείο 6 μετά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, έχουμε ένα συνάδελφο, τον Ερή και Σάμπον, που κατήγηλε το ότι δεν έλαβε εγκαίρως ε, την απάντηση από το Συμβούλιο για στα, στα ε, εμπρόθεσμα μετά από γραπτή ερώτηση και η Μπάρμπαρα Σπινέλη ε, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα σε μια ερχόμενη συνεδρίαση Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή οι γραπτέ ερωτήσει που υποβάλλονται και η καθυστέρηση απαντήσει. και θα πρέπει να προσεγγίσουμε όχι ειδικά αλλά γενικότερα το ζήτημα και γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση με τους συντονιστές μετά για προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα θυμάστε ότι κάναμε την ακρόαση τον Απρίλιο με ε, ευρύτατη συμμετοχή από όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Κάναμε τι διαπραγματεύσει και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την ε, για τα πεπραγμένα, για τις τελευταίες εξελίξεις και για την άποψή της σχετικά με το πώς μπορούμε με επιτυχία να ε, διεκπαιρεώσουμε αυτή τη διαδικασία προσχώρησης. Ενδεχομένως ε, προφορική ερώτηση με συζήτηση στην Ολομέλεια. θα ζητήσουμε από την Επιτροπή πρώτα να το συζητήσουμε μαζί μας και θα κρίνουμε πώς πρέπει να κινηθούμε μετά. Ε, Υπάρχει μια μελέτη από τον καθηγητή Ζάκε, θα ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα από το EPRS και την υπηρεσία τεκμηρίωσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου και ε, θα αφορά αυτό το θέμα προσχώρηση Ευρωπαϊκής Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατόπιν, επιστολή του Προέδρου Σούλτς ε, για την ε, επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς Για το, ε, την πολιτική ομάδα Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία. Αυτό είναι, αυτή είναι η επίσημη ονομασία και γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Σχετίζεται αυτό το θέμα με το ενδεχόμενο χρηματοδότηση και την ουσιαστική χρηματοδότηση αυτού του κόμματος από ε, τον προπολογισμό της Ένωσης. Ζητήσαμε λοιπόν γραπτή γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία και ε, από αυτή τη βάση στην επόμενη σύσκεψη των συντονιστών θα συζητήσουμε την έκθεση της ΑΦΚΟ για αυτό το ζήτημα και ε, θα συζητήσουμε το ζήτημα της ενεργοποίησης της διαδικασίας. Αυτές ήταν οι αποφάσεις των συντονιστών. Αν δεν ζητάει κάποιος το λόγο, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα οραμών. Πρόεδρε, άκουσα ότι η συνάντηση των συντονιστών συζήτησε το ενδεχόμενο να κληθεί ο κύριος Τίμερμανς για την πρωτοβουλία των πολιτών. Να σας ότι αυτό το δικαίωμα, ε, όσοι ασχολούνται με το δικαίωμα ε, έρευνας, ασχολούνται και με αυτό και ενδιαφέρονται για, αυτή την, για μια τέτοια ενδεχόμενη συνάντηση. Στην πρόσκλησή μου θα κάνω ε, ένα μακρύτερο κατάλογο θεμάτων, όχι μόνο αυτό που είπατε. Φυσικά απόκειται σε εσά. Από ό,τι θυμάστε, ο αντιπρόεδρος μας δεν ετοιμάζει γενικά ομιλίες, ε, σας ζητάει να υποβάλλετε ερωτήσεις. Μπορείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Υπάρχει και ένας μακρύς κατάλογος ούτως ή άλλως θεμάτων. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και καλό θα ήταν λοιπόν να μας δώσει κάποιες σκέψεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Τίμεν μας. Καθώς και για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας ε, της Κομισιόν, όχι μόνο για το τι συμβαίνει τώρα ή στο παρελθόν, αλλά και το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας. Καλό θα ήταν να μας μιλήσει και γι' αυτό ο κ. Μετά θα πάμε στο σημείο 5. Πάμε στο σημείο 5 που είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Έχουμε τα πρακτικά για τη συνεδρίαση της 22ης και 23 Φεβρουαρίου. Έχουν μοιραστεί τα πρακτικά και με βάση τη συνηθισμένη πρακτική θεωρούνται εγκεκριμένα αν δεν υπάρχει αντίρρηση η οποία θα υποβληθεί μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Υπάρχει τώρα το σημείο 6 στην ατζέντα, που όπως είπαμε δεν θα το συζητήσουμε. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε στην πραγματικότητα πριν από την προβλεπόμενη ώρα, που είναι 4.30. Άρα έχουμε άλλα 10 λεφτά στη διάθεσή μας. Άλλα 10 λεφτά για να ψυχαγωγηθείτε. Με οποιοδήποτε τρόπο σκεφτείτε. Αλλιώ πέστε μα κάτι. Ο Τζόρτζ, δεν θέλω να κάνω μια μακριά παρουσίαση. Να σε πιστήσω την προσοχή ε, στο ότι εγώ μπροστά μου έχω ένα έγγραφο που λέει 16 και 40, ότι 16 και 40 αρχίζει η ψηφοφορία. Άρα έχουμε 20 λεφτά, όχι 10 λεφτά. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, σταματήστε τα πηγαδάκια. Εσείς μπορεί να μην καταλαβαίνετε, αλλά γενικά δημιουργείται θόρυβος και δεν ακούμε. Ίσως να κάνω λάθος, αλλά για αυτό το σε αυτό το έγγραφο λέει ότι ξεκινάμε τις ε, ψηφοφορίες στις 16 και 40. Είπατε 16 και 30. Αν όμως έχουμε 20 λεπτά θα μπορούσαμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 8. Δεν έχουμε χρόνο. Ο Κρίστιαν Πρέντα δεν είναι εδώ, η Σιλβί Κάουφμαν δεν είναι εδώ, ο Μάικ δεν είναι εδώ ε, και δεν θα έρθει. Ή Μάικ. Και ο Κώστας δεν είναι εδώ. Μπάρμπαρα θα έρθει ή όχι. Δεν μπορούμε. Ο Φάμπιο, τέσσερις. Έχουμε τέσσερι και όδου εισηγητέ που λείπουν. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε το σημείο 8. Εντάξει. Έχω ένα έγγραφο από τον κύριο Πρέντα, εγώ πάντω, που μου έχει διαβιβάσει για να το αντικαταστήσω. Λόγω αυτού του λάθου πάντω, ο ενδεικτικό χρόνο ήταν 16 και 40. Πάντω, τα άλλα μέλη του ΕΛΚ θα φτάνουν όπου να είναι. Και μην ξεχνάτε ότι πολλοί ευρωβουλευτέ του ΕΛΚ είναι στο Λουξεμβούργο. Και δεν ξέρω λοιπόν πόσοι θα μπορέσουν να έρθουν. Καταλαβαίνετε που το πάω. No, we have the voting at 4.30 and then... Όχι, αμέσως μετά την ψηφοφορία που θα αρχίσει στις 4.30 θα συζητήσουμε αυτό το σημείο, το σημείο 8 δηλαδή. Συνάδελφοι, ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι νομίζαν τελικά ότι η ψηφοφορία έρχεται στις 16 ε, και 40. Ε, μόνο εγώ νομίζω, νόμιζα στις 16 ε, και 30. Έχουμε λοιπόν άλλα 15 λεπτά, θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε ας μιλήσουμε για το σημείο 9. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ είναι εδώ. Να σας πω που βρισκόμαστε με τη Διαθεσμική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες του follow-up και την ερμηνεία και εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Θα θυμάστε ίσως ότι η ΑΦΚΟ ε, πρέπει να ετοιμάσει μια γνωμοδότηση, τη ζητήθηκε να ετοιμάσει μια γνωμοδότηση που θα αναλύει και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης Και επίσης ε, θα πρέπει ε, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου να του ζητήσει ε, του πρόεδρου του Κοινοβουλίου να υπογράψει εκ μέρου του Κοινοβουλίου τη συμφωνία για το Better Lawmaking. Στις 9 Μαρτίου το αναφέραμε στην Ολομέλεια, το θέμα αυτό της έκθεσης και συνεχεία το θέμα αυτό το συζητήσαμε και η ΑΦΚΟ και η Γιούρη ανεξάρτητα οι δύο επιτροπές, για το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία εφαρμογής αυτής της διαθεσμικής συμφωνίας. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια κοινή ομάδα εργασίας, γιατί η έκθεση για την εφαρμογή υπόκειται στο άρθρο 55 και ετοιμάζεται από δύο επιτροπές, την ΑΦΚΟ και την Επιτροπή Γιούρι. Σταγματικών και νομικών υποθέσεων. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή την κοινή ομάδα εργασίας για να διευκολύνουμε τη διαδικασία συνεργασίας ούτως ώστε να μην πρέπει κάθε φορά να συγκαλέσουμε και τις δύο επιτροπές χώρια, αλλά να είμαστε πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί μέσω της ομάδας αυτής εργασίας. Έχει ήδη συνεδριάσει μια φορά η ομάδα εργασίας και συμφωνήσαμε ότι θα είναι και μια πλατφόρμα διευκόλυνσης των δύο εισηγητών, του Richard Κόμπερ του ΑΦΚΟ και του εισηγητή της Γιούρη, που χρειάζονται μια πλατφόρμα για να συζητούν θέματα. Υπάρχει βεβαίω πλατφόρμα η ομάδα εργασία, αλλά η ομάδα εργασία παρακολουθεί και την αρχική εφαρμογή τη διαθεσμική συμφωνία. Χρειάζεται όμω και μια πλατφόρμα, ούτω ώστε όλε οι άλλε επιτροπέ οι οποίε θέλουν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή, στη διαδικασία εφαρμογή να μπορούν και αυτέ να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Μπορούν λοιπόν να έρχονται στην ομάδα εργασίας και να συζητάνε τα θέματα εκεί. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου συγκάλεσε και μια ομάδα, την ομάδα των τεσσάρων. Η ομάδα των έξι ήταν για την Κίνα. Όχι, γιατί τέσσερι ήταν και εκεί. Άλλη μια ομάδα τεσσάρων λοιπόν. Ο, ο κύριος Φερχόφστατ, οι δύο εισηγητές, ο, ο κύριος Κόρμπερ και ο εισηγητής της Γιούρη, που είναι και πρόεδρος της Γιούρη, και εγώ, έχουμε δύο πρόεδρους δηλαδή, που θα βοηθήσουμε στην ομάδα εργασίας. Ο Κώστας Φόμπονταρ, Χιούμπνερ και Κόρμπετ είναι στην ομάδα των τεσσάρων. Θα συνάψουμε κοινά συμπεράσματα, θα τα προτείνουμε στην διάσκεψη των Προέδρων για να δώσουμε μία πρόταση για το πώς θα προχωρήσουμε με την φάση του follow-up της συμφωνίας. Θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Όσοι είστε στην ίντα ή στην ΑΦΕΤ θα ξέρετε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ και μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για, τη, για όλες τις διεθνείς συμφωνίες όπου προτείνουμε ότι η ΑΦΕΤ και η ΙΝΤΑ θα είναι καθήλυνα αρμόδιε επιτροπέ για τι διαπραγματεύσει, αλλά υπάρχουν και διαπραγματεύσεις ούτω ώστε να καθοριστούν κριτήρια για την, ε, τις εκτελεστικές και κατεξιοδότηση πράξης και όσοι ασχολείστε με τα νομοθετικά θέματα ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Η βασική αλλαγή που είναι σημαντική για μας είναι η αλλαγή για την οποία είναι υπεύθυνος ο Ρίτσαρντ. να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση δηλαδή ανάμεσα στον εσωτερικό κανονισμό του Rules of Procedure που είναι σε φάση προετοιμασίας και μεταρρύθμισης με την διαθεσμική συμφωνία. Είναι πολυεπίπεδη δουλειά αυτή που μας περιμένει. Μέσα από, τα, από τις ομάδες που έχουμε και τις δομές που έχουμε θα τα καταφέρουμε. Και σύντο χρόνο πιστεύουμε ότι οι δομές αυτές θα γίνουν λιγότερο μπαρόκ και πιο μοντέρνες και απλές, εάν τα πράγματα πάνε κατευχή. Ο Ρίτσαρτ λοιπόν και εγώ ασχολούμαστε με το follow-up, με τη συνέχεια που θα δοθεί στη διαθεσμική συμφωνία και θα εξασφαλίσουμε και την ευθυγράμμιση. Εδώ έχουμε φτάσει με τη διαθεσμική συμφωνία. Φαντάζεστε επίσης και τις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές που θα πρέπει να γίνουν και την, ε, η εφαρμογή της έκθεσης είναι σημαντικό πράγμα, αλλά είναι ένα πράγμα. Το άλλο είναι ότι όλες οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου εμπλέκονται πάρα πολύ στο θέμα της συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα και στη διαδικασία της βελτίωσης νομοθετικής προσπάθειας. Έχουμε και τους εκπροσώπους της Διαθεσμικής Συντονιστικής Ομάδας με την κυρία Φραντσέσκα Ράτη και από την διοίκηση υπάρχει και ένα project team που συνεργάζεται μαζί μας επίσης. Υπάρχει πολλοί κόσμος λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον και από την πλευρά του, της διοίκησης του Κοινοβουλίου. Όλα τα θεσμικά όργανα τώρα προσαρμόζονται εσωτερικά δουλεύουν διαφορετικά για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα συμφωνία. Και ακριβώς θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τίμερμανς τι μπορεί να μας πει ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διευκολύνουμε και όχι θα δυσκολεύσουμε τη συνεργασία. Θα είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να συναντηθούμε τον κύριο Τίμερμανς για να του θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό είναι το σημείο 9 στη μέση διάταξη. Επίσης συμφωνήσαμε ότι θα σας ενημερώσουμε τακτικά, θα σε ενημερώνουμε τακτικά για τη δουλειά της ομάδας εργασίας και ο Ρίτσαρντ ούτως ή άλλως θα έρχεται εδώ και θα μιλάει για την έκθεση. Αυτή η διαθεσμική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθετικής προσπάθειας δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει μπει ας στο, στο ντουλάπι. Είναι κάτι το οποίο ε, μεταμορφώνεται, αλλάζει μέρα με τη μέρα και θα σας ενημερώνουμε σύντο χρόνο. Ο Χέλμου Σόλτ θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ παρά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία γιατί σίγουρα αυτή η εργασία περιλαμβάνει διάφορους τομείς. Θα ήθελα να ξέρω η ομάδα αυτή εργασίας πώς ε, συνεργάζεται με άλλα όργανα τα οποία έτσι και λιώς έχουν κάποια επεξεργασία και κάποια εμπλοκή στις ε, διεθνείς συμφωνίες. Θα ήθελα να καταλάβω πώς ε, δομικά, διαρθρωτικά συνδέονται αυτή η ομάδα εργασίας με τα υπάρχοντα όργανα στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχει διαφάνεια. Να κατανοήσουμε κι εμείς, αλλά βεβαίως να είναι και πιο αποτελεσματική η εργασία αυτών και εμείς οι μεμονωμένοι ευρωβουλευτές να μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστώ. Ρίτσαρτ, ένα λεπτό να απαντήσω. Ναι, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας προανέφερα δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικά πολλούς ρόλους, όπως σας το παρουσίασα προηγουμένως. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, χάρη στην κοινή γραμματεία και στο άρθρο 55, δηλαδή οι δύο επιτροπές επί ίσης εργάζονται, και επειδή ακριβώς προετοιμάζεται ένας κατάλογος θεμάτων, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για αυτές τις δύο οργανικές συμφωνίες, και επειδή υπάρχουν και διάφορα επίπεδα όσον αφορά τον επίγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, μια ιεράρχηση, παραδείγματο χάρη τον Ιανουάριο, υπήρχε μια ιεράρχηση των θεμάτων και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ο Ρίτσαρτ έτσι κι αλλιώ έχει ήδη παίξει το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ ημών και των άλλων θεσμικών οργάνων και σαφώς και οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν για την εργασία στο εσωτερικό αυτής της ομάδας εργασίας είναι πολύ σαφείς. Δεν υπάρχει πάντως, ε, αν θέλετε, απόσταση ή διαφορές μεταξύ αυτών που αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε πρόκειται για την ομάδα εργασίας είτε πρόκειται για τα άλλα όργανα. Και αυτό διότι διέπεται η εργασία όλων μας από τους ίδιους κανόνες. Και ουσιαστικά αυτή η ομαδική εργασία γίνεται με την βοήθεια της γραμματείας όπως σας είπα, η οποία μας ενημερώνει, μας δίνει και κάποιες πολιτικές ε, κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Αυτή η ομάδα εργασίας δεν διευκολύνει απλώς τη συνεργασία των δύο επιτροπών, αλλά διασφαλίζει τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζονται για αυτά τα θέματα. Ξέρετε πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις διάφορες υπηρεσίες. Βεβαίως, ο ρόλος αυτής της ομάδας εργασίας είναι καθοριστικός και πρέπει κάθε φορά να ενημερώνονται οι επιτροπές. Θα ενημερώνουμε εδώ την ε, δική μας επιτροπή, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα η οποία θα διασφαλίσει την συνάφεια της επεξεργασίας μεταξύ των διαφόρων ε, οργάνων και ομάδων. Ρίτσαρτ, θες να προσθέσεις κάτι? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση του κύριου Σόλτς και εξαιρετική και η απάντηση που έδωσες. Αυτά. Ανησυχούσαμε ότι θα μπορούσε ουσιαστικά να χαθεί ο στόχος, γιατί βεβαίως υπάρχει η διάσκεψη των προέδρων, η διάσκεψη των κεφαλής των επιτροπών, των πρόεδρων των επιτροπών. Πολλές είναι, αν θέλεις, οι υπηρεσίες που εμπλέκονται και οι επιτροπές. Και όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, βεβαίως τα θέματα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομοθετικά θέματα, η επιλογή της διάσκεψης προέδρων είναι πολύ σημαντική εδώ. Αλλά βεβαίως και η Επιτροπή ΑΦΕΤ, η Επιτροπή εμπορίου σίγουρα έχουν ε, πολύ αυξημένο ενδιαφέρον. Οι περισσότερες πιστεύω επιτροπές θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία σε κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι για πρώτη φορά Είναι η δεύτερη διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία που παρακολουθώ, στην οποία εμπλέκομαι και θεωρώ ότι αυτή τη φορά εμπλέκονται πολύ καλύτερα και συμμετέχουν με πολύ πιο ενεργό τρόπο οι διάφορες επιτροπές μέσω αυτής της νέας δομής. Μπορούμε νομίζω, αν κανείς δεν ζητάει το λόγο, αν κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο, μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Είναι η ώρα των ψηφοφοριών. Ναι. We have to Μπορείτε να ελέγξετε ότι λειτουργεί το σύστημα. Δοκιμάστε τις κάρτες σας. Αρχή της α, ψηφοφορίας ελέγχουμε. Ε, Εντάξει. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Πρόκειται για το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο, νομοδότηση, συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, ελέγχουμε, τροπολογία 1, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά. Νομίζω απορρίπτεται η 4. Συμβαστική Β υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 δεύτερο τμήμα Οκτώ δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται, ελέγχουμε την 8 δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 δεύτερο τμήμα υπέρ 15 δεύτερο τμήμα κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία το δεύτερο της 15 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Απορρίπτεται. 10... 18. 18, τροπολογία 18, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Αφού δεν θέλετε να ελέγξουμε, δεν ελέγχουμε, εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά ελέγχουμε 29. Αρχή της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 29. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται 14 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Μπράβο. ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώσαμε και τις ψηφοφορίες. Και περνάμε τώρα στο σημείο του κυρίου Άνεμανς. Πρόκειται για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ετήσια έκθεση του 2014. Σας δίνω το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, σας παρουσιάσω την έκθεση σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής ε, του δικαίου της Ένωσης. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την έκθεση Χάουταλα. Τοποθετήθηκα για όχι γενικά, δηλαδή για τη στάση των ε, ε, θεσμικών οργάνων, αλλά παρέθνησα μόνο τα γεγονότα και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε. Είμαι πολύ συγκεκριμένο ε, μέσα στη γνωμοδότηση και θα είμαι σύντομο στην παρουσίασή μου. Για την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, αυτό είναι το βασικό θέμα που με απασχολεί. μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι μειώθηκε ο ρυθμός των διαδικασιών 265 καθώς και τα προδικαστικά ερωτήματα. Ε, η κυρία Χαουταλά θεωρεί ότι ε, για τα, στο τωρινό πλαίσιο και με την τωρινή κατάσταση των πραγματών τα κράτη-μέλη θα ήταν καλό να ε, κινούν τις διαδικασίες για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θέλαμε να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην ε, διαφάνεια. Ανέφερα επίσης ότι ως προς τις σχέσεις ε, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει να επικρατήσει διαφάνεια. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Δεν θέλω και να προσθέσω πολλά πράγματα, υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτο μου ζήτησε να διαβάσω τα εξή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άνιμανς ε, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, αλλά ξέχασε ότι κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά εφαρμόζει τις συνθήκες σε βάση του άρθρου 17 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να θυμίσουμε στον κύριο Άνεμενς είναι ότι όταν ένα κράτος μελός δεν τηρεί κάποια προθεσμία για τη μεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό συνιστά παραβίαση των συνθήκων και θα πρέπει να τύχει ε, της ανάλογης μεταχείρισης. Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε σχέση με το ότι είναι, αποτελεί προϋπόθεση η σωστή εφαρμογή του δικαίου για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Φαίνεται ότι είναι όλα τέλεια αν διαβάσει κανείς την έκθεση του κυρίου Άνμανς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως. Ε, Ότω καλωσορίζουμε τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάση, καθώς και τι προσπάθειε που κάνουν τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με, το, με την κειμένη νομοθεσία. Όμως, ταυτόχρονα να απευθύνουμε έκκληση ε, προς, τα κράτη-μέλη για εγρήγορση σε σχέση με την μεταφορά, διότι η ε, εσφαλμένη μεταφορά πλήττει κυρίω του πολίτε. Ε, το 2014 βλέπουμε στην αντίστοιχη έκθεση ότι ε, παραμένει πρόβλημα η καθυστέρηση ως προς τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των οδηγίων. Θα ήθελα να τονίσω και κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Η Επιτροπή έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες για να αναπτύξει μέτρα για την πρόθεση της συμμόρφωσης ε, σε γιατί έχουμε το 75% του ποσοστού εφαρμογής του ποσοστού EU Pilot. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες με την νέα δικτυακή πύλη για την εφαρμογή του δικαίου. Είναι σημαντικό για τα κράτη-μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τους πίνακες συσχετισμού με, ε, ε με ξεκάθαρες πληροφορίες όπως αυτό προβλέπεται. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε την, ε, την υπερβολική, τις υπερβολικές ρυθμίσεις ε, ως προς την μεταφορά του δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Αυτό προβλέπεται στο Better Lawmaking, στη νέα διοργανική συμφωνία που διέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων. Δεν είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα και ε, οι ευρωσκεπτικιστέ υποφελούνται όταν υπάρχει ασφαλμένη εντύπωση σε σχέση με ε, τα όσα ισχύουν για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, ήθελα να στήσει και παράταση ο κύριο Πέρατα με τι 6 ώρα ή δυνατόν. Θα, θα το σκεφτούμε. Θα το ελέγξει η γραμματεία και θα σα πούμε. Αλλά μα πιέζουμε κιόλα διότι έχουμε και την ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Εντάξει, 6 το απόγευμα δεν είναι υπερβολικό. Το οι σοσιαλιστές, η Σίλβια δεν είναι εδώ, οι Μερσέντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Κάουφμαν δεν μπορεί να παραστεί και μου άφησε ένα σύντομο σημείωμα. όπου ζητάει ότι δεν έχει να κάνει δικέ ή ιδιαίτερε παρατηρήσει στην έκθεση. Χαιρόμαστε που υπάρχει μία μείωση των παραβιάσεων ούτως ή άλλως των ευρωπαϊκών κανόνων, παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι ρόδινα και έχουν επιληθεί όλα τα προβλήματα. Πάντως, είναι σημαντικό να μας ξεκαθαρίσει η Κομισιόν, εξηγώντας μας σε τι φάση εφαρμογής ε, βρίσκονται τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμφωνούμε επίσης ότι αν υπάρχουν παρατηρήσεις, καλό είναι να γίνονται εκ των προτέρων, παρά να μην εφαρμόζουν τα κρατη την νομοθεσία γιατί ξέχασαν να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις ή να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις που, ή κάποια θέματα ας πούμε, που δεν τους ικανοποιούν ή που δεν τα θεωρούν σωστά ή δεν συνάδουμε τη δική τους θεώρηση για την Ευρώπη. Να τις κάνουν λοιπόν τις ερωτήσει και τις πατήσεις πριν και να μην καθυστερούν την εφαρμογή. Τώρα, δεν έχουμε παρατηρήσεις. Εμείς θα αξιολογήσουμε το αν χρειάζεται να υποβάλουμε τροπολογίες και με βάση την τελική έκθεση θα εκφράσουμε μία γνώμη και θα λάβουμε υπόψη βεβαίω και τις τροπολογίες που θα παρουσιαστούν και θα εγκριθούν από το ECR. Θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, συνάδελφοι. Υποστηρίζω πλήρως την, την εκνομοδότηση που παρουσίασε ο συνάδελφος. Πιστεύω ότι είναι ευσύνοπτο έγγραφο υποστηρίζει και τον βασικό στόχο που είναι η πιο έγκαιρη ε, εφαρμογή του, των ε, οδηγιών του δευτερογενούς δικαίου, διότι γι' αυτό μιλάμε. Επίσης, τονίζει την αρχή της επικουρικότητας, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να πριτανεύει και σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα, όπως και τα υπόλοιπα θέματα, θα πρέπει να συζητούνται με βάση τα εξής. Το κλειδί για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη, μεταξύ δηλαδή των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χαιρόμαστε για την γνωμοδότηση που μόλις λάβαμε και που μοιάζει να διέπεται από αυτές τις αρχές. Δηλαδή να υποστηρίζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της περαιτέρω ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμπιστοσύνη, λοιπόν, Σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, στο έγγραφο. Από τους φιλελεύθερους υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει. Μάιτι. Από, τους, ε, από την ΚΟΕ υπάρχει κανείς και από την EFTD ουδής. Τελικά δεν είναι μόνο το ΕΛΚ που γιορτάζει στο Λουξεμβούργο, όλοι κάπου αλλού βρίσκονται. Ευτυχώ η προθεσμία δεν είναι αύριο, αλλά μεθαύριο. Έξι όμως το απόγευμα. 1η Ιουνίου, 6 το απόγευμα. Εν συνεχεία ψηφίζουμε στις 15 Ιουνίου, λόγω της προφορίας στην Επιτροπή Γιούρη, της αρχές Ιουλίου. Άρα, κύριε Άνεμανς, Κάρολ, θέλετε να μιλήσετε? Όχι, όχι. Θα διαβάσω με ναι. μεγάλη προσοχή. Θα διαβάσω με μεγάλη προσοχή τις τροπολογίες που θα υποβάλουν ε, ενδεχομένω οι συνάδελφοι. Δεν έχω πάντως κάτι να προσθέσω. Δεν είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής στην αίθουσα. Θέλετε κάτι να πείτε στα πλαίσια αυτών που ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μάριος Ντάτσα και είμαι από την ε, υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Με μεγάλη προσοχή διαβάσαμε τις προτάσεις ε, του εισηγητή. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις ε, της Επιτροπής σίγουρα θα συνεισφέρουν σε μια πολύ πιο έγκαιρη επίλυση των υποθέσεων ε, διαδικασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει σαν διαδικασίες επί παραβάση και βεβαίως η καθυστερημένη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο είναι αυτό που συνήθως ε, μας προβληματίζει. Εμείς ε, βεβαίως και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν εγκαίρως τις ε, οδηγίες και την υπόλοιπη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό τους δίκαιο. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και μία πληροφόρηση από μέρους των κρατών μελών όσον αφορά την υιοθέτηση των ε, νομοθετικών κειμένων και αυτό να γίνεται σε πρώτα στάδια της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε αυτή την ενημέρωση γιατί μας βοηθάει να βελτιώσουμε τα μελλοντικά κείμενα της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σημείο έχει μείνει στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώσεις που αφορούν την επόμενη συνεδρίασή μας. Στις 15 Ιουνίου θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση. 9 με 12.30 και το απόγευμα. Θα συναντηθούμε λοιπόν στις 15 Ιουνίου. Τέλος της συνεδρίας.